Buongiorno a tutti, cominciamo. vi Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν καλό θα είναι να έχετε μαζί τις ε, <coughs> για την ψηφοφορία μετά. Ε, η ακρόαση του κυρίου Εκβίλτα αναβλήθηκε. Θα ορίσουμε αργότερα σήμερα πότε θα γίνει. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι ο διορισμός ενός νέου μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κύριος Χάγκαρντ Χόγκερμπάουερ. Ορίστηκε ως υποψήφιος από τις Αυστριακές Αρχές. Τον καλωσορίζω και του δίνω και το λόγο για μια σύντομη αυτοπαρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα την ευκαιρία να ε, συστηθώ ενώπιόν σας και πάρα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου ως προς την μεταξέλιξη του ελέγχου των οικονομικών στην Ευρώπη. Εγώ γεννήθηκα στη Βιέννη, ε, πήγα και στο γυμνάσιο στην ε, Ακαδημία τη Θηρεσιανή, με τέσσερις ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια ε, περί απτυχίο έκανα τη στρατιωτική μου θητεία. Κατά τη διάρκεια ε, των επιστημών μου, το των σπουδών μου, συγγνώμη, όταν σπούδαζα νομική, ε, και οικονομικά. Σε ηλικία 21 ετών πήρα το διδακτορικό μου. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη τύχη, διότι ε, στην Αυστρία δεν παίρνει κατευθείαν από το πανεπιστήμιο στο ελεγκτικό συνέδριο, γιατί περιμένουν εμπειρία και επαγγελματική ε, πείρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή τόσο γρήγορα πήρα διδακτορικό, με πήρα μέσα ο διευθυντή του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ηλικία 21 ετών. Στη συνέχεια στο Ελεκτικό Συνέδριο της Αυστρίας. Ε, ήλεγχα επί μία πενταετία ε, ε οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης και ε, ασφάλιση ατυχημάτων. Στη συνέχεια ε, μου ζήτησα να πάω στο κοινοβούλιο και να αξιοποιήσουν εκεί και πολιτικά την εμπειρία μου από το ελεγκτικό συνέδριο. Παρ' όλα αυτά παραμένω μέχρι και σήμερα υπάλληλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή από το 1974 ε, η οργανική μου θέση είναι στο ελεγκτικό συνέδριο. Αργότερα έγινα και υπάλληλο ε, της διεύθυνσης της Βουλής. Γι' αυτό λοιπόν από το 79 που σας είπα Έφυγα από το ελεκτικό συνέδριο και πήγα στη Βουλή γιατί διαπίστωσα κατά τη διάρκεια των εργασιών μου ότι πολλά από αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, αλλιώς δεν εφαρμόζονται. Και εκεί σκέφτηκα ότι μπορώ ενδεχομένω με βάση ε, την εμπειρία μου στην ελεκτική διαδικασία να εφαρμόσω και με τη βοήθεια της πολιτικής κάποια πράγματα στην πράξη. Αυτό εν μέρη το κατάφερα, βέβαια δεν τα πετυχαίνει κανείς πάντα όλα, είναι σαφές αυτό στο Κοινοβούλιο ε, ε, έδινα συμβουλές ε, στην Επιτροπή Ελέγχων των Λογαριασμών. Δηλαδή είχα διπλή ιδιότητα. Ως ελεγκτής συνεργαζόμουν με το Κοινοβούλιο και ε, από πλευρά τη Βουλή ήμουν ε, ο σύνδεσμο, αν θέλετε, ε, τη αρμόδια επιτροπή με το ελεκτικό συνέδριο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για να υπάρχει και απρόσκοπτη συνεργασία. Εκτό από το, την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, συμβούλευα και άλλες επιτροπές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Πάντα στην Αυστριακή Βουλή. Ταυτόχρονα και παράλληλα είχα και κάποιες ε, πολιτικές θέσεις, ε, ε, πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σύμβουλος διαφόρων οργανισμών και για άτομα με αναπηρίες και για κοινωνικές υποθέσεις. Είχα λοιπόν πολλαπλές δραστηριότητες που πάντα προϋπόθεταν ανεξαρτησία, όχι μόνο Ε, ε, και είχα και αποπτικές δραστηριότητες και ε, ας πούμε στη διανομή, όχι ακριβώς διανομή των, των αδειών για την ελεύθερη ραδιοφωνία, την ιδιωτική ραδιοφωνία. Εντάξει, μοίραζα εγώ τις άδειε, αλλά συμμετείχα σε αυτό το όργανο και στο Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως σας είπα, διατέλεσα πρόεδρος επί σειρά ετών στην αρχή ήταν ένα πολύ επίμαχο όργανο αυτό και οι ψηφοφορίες γινόντουσαν σε κλίμα τεταμένο με κομματικά κριτήρια. Από τότε που ανέλαβα εγώ πρόεδρος τα πάντα προχωρούσαν συνενετικά και ε, γνωρίζω πολύ καλά πώς να διατηρώ την ανεξαρτησία μου. Επίσης ήταν πάντα σημαντικό για μένα να έχω υπόψη μου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αδιαδρομία μου παρέμενα και υπάλληλο του ελεγκτικού συνεδρίου και υπάλληλο της Βουλής. Και αυτό μου έδινε ανεξαρτησία στις δραστηριότητες μου, τις υπόλοιπε. Ε, γιατί υπέβαλα τώρα υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για μένα είναι σαφέστατο αυτό. Η σημασία του προϋπολογισμού ε, και του των οικονομικών στην Ένωση είναι όλο και πιο σημαντική, πιο μεγάλη και επίσης οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι ε, τα χρήματά τους την χάνουν σωστής διαχείρισης και, και φρόνιμης διαχείρισης για να αρθούν ε, κάποιες ε, επιφυλάξεις και κάποιες αμφισβητήσεις που κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Το λόγο στην συνάδελφα Γιάλα, η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βέγκερ Μπάουερ στην Επιτροπή μας ως υποψήφιο που προτείνει η Αυστριακή Κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορείτε να μας διευκρινίσετε ορισμένα στοιχεία, τα οποία έχετε απαντήσει βεβαίω ορισμένα γραπτός, αλλά κάποια άλλα όχι. Και νομίζω θα μπορούσε να μας βοηθήσει η προφορική σας απάντηση, ε, διευκρινιστικά. Σε ό,τι φορά το βιογραφικό σας, λέτε, και είναι ενδιαφέρον αυτό, ότι ήσασταν υπάλληλο του ελεγκτικού συνεδρίου και θεωρήσατε ε, δεδομένης της ε, εμπειρίας σας στον έλεγχο των λογαριασμών που συνδέεται αυτό με τις πολιτικές αποφάσεις, θεωρήσατε σκόπιμο ε, να ε, προχωρήσετε και στην πολιτική για να βοηθήσετε. Και το 79 μας λέτε, ή λίγο αργότερα, εμφανίζεστε ως ε, πολιτικός διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό πώς γίνεται. Γιατί όπως και εσείς ο ίδιος είπατε, βασικό στοιχείο είναι ανεξαρτησία. Όχι μόνο από το κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται ο ελεγκτής, αλλά και η ικανότητα ανεξαρτησίας και ιδιότητα ανεξαρτησίας από κομματικά, ε, κομματικούς δεσμούς. Μας είπατε ότι πετύχατε ορισμένα πράγματα, όχι όλα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για ε, το τι δεν καταφέρατε να ε, πετύχετε ε, από πλευράς κοινοβουλευτική και τι είχε προταθεί. Πολιτικά ε, ρωτώ. Και κάτι άλλο τώρα. Σας ρωτήσαμε εάν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας χρειάστηκε να κάνετε λογιστικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο Μα είπατε ότι στην Αυστρία δεν γίνεται τέτοιο έλεγχο. Είναι η ερώτηση υπαριθμό 4 που σα έχει υποβληθεί. Ωστόσο, λίγο παρακάτω, ε, λεπτομερώς εξηγείται πώ εγκρίνεται στην Αυστρία η εκτέλεση του προπολογισμού και διαχείριση ε, και ε, ότι συμμετείχατε στην αυτή δημοσιονομική διαχείριση των έλεγχων. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μετάφραση. Μήπω μπορούσατε να μα διευκρινίσετε αυτή την αντιστοιχεία. Και επειδή πάντα κάνουμε λίγο μια επαλήτηθευση των στοιχείων για να αξιολογήσουμε τον υποψήφιο, το 2008 κυκλοφόρησε σε κάτι δημοσιεύματα στον τύπο ότι ο ρόλος σας στο Συμβούλιο Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων ως Διευθυντής ή Πρόεδρος που διατελέσατε εκεί ε, συνδέθηκε με κάποιες επικρίσεις ότι μέσω τροπολογίας δεχθήκατε ε, να αρχίσει η παρακολούθηση των διευθύνσεων IP, των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στο διαδίκτυο, χωρίς προηγούμενη δικαστική εντολή ή άδεια για να μπορέσει κανείς να παρακολουθεί και να ερευνά τις ε, διευθύνσεις ε, των χρηστών του διαδικτύου. Γι' αυτό εσείς τι λέτε γιατί ό,τι έχει να κάνει με προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων για μας θεμελιώδες. Επίσης σας έχουν κατηγορήσει ότι περιορίσατε τις συνεδριάσεις ε, ε, από 8, το, το, του Συμβουλίου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων, από 8 που ήταν αρχικά τις περιορίσατε, τις μειώσατε σε 5. Ένα, κανονικά λέτε ότι καλύτερα, μάλλον κάπου αλλού ε, ισχυρίζεται ότι για να υπάρχει καλύτερος έλεγχο, χρειάζεται τα ελεκτικά συνέδρια να συνεδριάζουν πιο συχνά. Στη δική σας χώρα όμως κάνετε το αντίθετο. Αυτά, Πρόεδρε, είχα ω ερωτήσεις και στη συνέχεια θέλω να επεκταθώ και επί τη ουσία. Ευχαριστώ. Grazie. Äh, μάλιστα. Πολιτικός διευθυντής σε εμάς τι σημαίνει. Ότι ήμουν αρμόδιος για την διοργάνωση των επαφών μεταξύ της πολιτικής ομάδας, ε, της, του κυβερνητικού κόμματος, ε, και του Ομοσπονδιακού Κόμματος και των τοπικών. Σε διοικητικό επίπεδο δηλαδή των τοπικών περιφερειακών οργανώσεων Ήμουν προσωπάρχης, αν θέλετε, ε, στη ε, πολιτική δουλειά ε, της πολιτικής μου ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαιρνα πολιτικές αποφάσεις εγώ. Τις προετοίμαζα και είχε τη δυνατότητα έτσι το κόμμα σε επίπεδο κυβέρνησης, βουλής, ε, ξέρετε ότι η Αυστρία είναι ομοσπονδιακή ε, δημοκρατία και έχει διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Ήταν λοιπόν πολιτικός βέβαια και σαφώ, αλλά γιατί είχα και αρμοδιότητες στο ιστορικό της ομάδας σχετικές με τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι μια δραστηριότητα διοικητική, πολιτικής διοίκησης, αλλά διοικητική. Η δεύτερη ερώτηση, ανεξαρτησία. Προσπάθησα πολύ σύντομα να σας το περιγράψω πάντα πρόσεχα ανέκαθεν να παραμένω υπάλληλο. Κυρίω υπάλληλο του ελεκτικού συνεδρίου και όπω σα είπα αργότερα έγινε και υπάλληλο ε, τη διεύθυνση τη Βουλή. Επί Alois Μοκ και συνεργάστηκα με το πιο στενό του συνεργάτη και ήταν και συντονιστής της ε, πολιτικής ομάδας και ήρθε και μου είπε ε, ότι δεν έχει νόημα να παραμείνω υπάλληλο του ελεγκτικού συνεδρίου, αφού έτσι κι αλλιώ είναι μόνιμη η θέση μου στην πολιτική ομάδα, στο κοινοβούλιο και μήπω θέλω να παραιτηθώ από το ελεκτικό συνέδριο, να παραιτηθώ από δημόσιο υπάλληλο γενικά. Εγώ του είπα ότι ποτέ αποκλείεται να παραιτηθώ από δημόσιο γιατί θέλω να διατηρήσω την ανεξαρτησία μου. Ο δόκτωρα Λοϊ Μοκ, προϊστάμενό μου, εξεπλάγει και είπε. Μα συνεννοούμαστε τόσο καλά, έχουμε τόσο καλές σχέσεις, δεν πρόκειται να σου συμβεί τίποτα. Και εγώ είπα όχι, θέλω να μπορώ να προχωρώ πάντα με ψηλά το κεφάλι χωρίς καμία εξάρτηση από οποιοδήποτε πολιτικό, ακόμα και από πολιτικό του ιδίου μου του κόμματο. Το επόμενο θέμα. Τι δεν πέτυχα από αυτά που φιλοδοξούσα. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα ε, κοινωνικής ασφάλισης, ε, συντάξεων, ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ατυχημάτων. Στον προπολογισμό αυτό είναι μεγάλο κονδύλι. Και έχουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα στις ασφάλειε των συντάξεων λόγω τη δημογραφική εξέλιξη. Αυτό το αντιμετωπίζουν σχεδόν όλε οι βιομηχανικέ χώρε και είναι βασικό πρόβλημα. Κάναμε μεγάλα βήματα στι αρχέ του 21ου αιώνα για την εξασφάλιση ε, των συντάξεων με μεγάλη συνταξιωτική μεταρρύθμιση. Έκτοτε όμως έχουν οπισθοδρομήσει όλο και περισσότερο και η εξασφάλιση των συντάξεων είναι κάτι το οποίο δεν έχει λυθεί τουλάχιστον στη χώρα μου γιατί η δημογραφική εξέλιξη είναι μη αντιστρεπτή και αν αλλάξει σήμερα κάτι για τις συντάξει έχει βάθος δεκαετιών μέχρι να αποδώσει. Γιατί ακόμα και μια πληθυσμιακή πολιτική δεν μπορούμε να την αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολύ ε, μεγάλη προσπάθεια. Αυτό λοιπόν το εργοτάξιο ε, είναι υπόθεση ετών και ομολογώ ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει αυτά που θα θέλαμε. Ακόμα και αν συμμετέχω σε ένα κόμμα που κυβερνάει, ε, πρέπει να σας πω ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν έχουμε επιτυχεί όσα θα έπρεπε. Και ένα δεύτερο, για να μην μακρηγορώ πολύ, είναι τα θέματα της υγείας, υγειονομικής περίθαλψης. Και εδώ το ίδιο πρόβλημα έχουμε, τη δημογραφική εξέλιξη. Ο κόσμος γερνάει, αυξάνονται οι απαιτήσει ε, για περίθαλψη και λόγω ιατρικής πρόοδου αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής και εδώ είναι ο άλλος μεγάλος τομέας, το μεγάλο κονδύλι που επιβαρύνει πολύ και τα δημόσια οικονομικά. Ούτε αυτό έχει λυθεί σε καμία περίπτωση ακόμα στην Αυστρία. Είναι μια διαδικασία μόνιμη εν εξελίξη. Αυτά τα δύο δεν τα απέτυχα όσο θα ήθελα. Για την έγκριση της δημοσιονομικής διαχείρισης. Είχα αρμοδιότητα, ε, ε, παρακολουθούσα και συμβούλευα ε, για κάποια θέματα, κεφάλαια του προϋπολογισμού, δηλαδή εργασία και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή, κατεθέτει τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο, και μετά πηγαίνει αυτή η πρόταση σε επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου και συζητούν σε λεπτομέρειες. Εκεί έκανα εγώ τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Για την απαλλαγή και τον έλεγχο των λογαριασμών, σε εμά γίνεται ως εξή. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, εκπονεί ε, μια πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Ε, μετά από πρόταση των Υπουργείων, ελέγχει αυτά που προτείνουν τα Υπουργεία και εκθέτει ε, εκδίδει την έκθεσή του με αξιολογήσεις και στατιστικές και οικονομικές. Δεν είναι μόνο λογιστική οι λογαριασμοί μας και η αντιμετώπιση μας, αλλά είναι και θεματική και τελικά... Ε, στην Επιτροπή του ελεγκτικού συνεδρίου διαβιβάζουμε αυτή την πρόταση για το κλείσιμο των οργανισμών ε, και την αξιολογεί είτε στο σύνολό του και στο σύνολό του και επί της αρχής και στα κεφάλαια. Και τελικά, σε περίπτωση που είναι θετική η αξιολόγηση και η απόφαση της Επιτροπής του Ελεκτικού Συνεδρίου, τότε και μόνο τότε πηγαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής. Και στην Ολομέλεια εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται. Και αυτή τη στιγμή εγκριθεί αυτή η έκθεση, απαλλάσσεται η κυβέρνηση. Τώρα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εσείς διαβάστε μόνο τις πράσινες εφημερίδες για αυτά που λέτε. Ομολογώ ότι στο Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, ε, αλλά άλλες φορές ήταν ομόφωνες με μία ψήφο κατά και η αντίθετη ψήφος ήταν των πρασίνων. Ε, ο εκπρόσωπός τους, ο Δόκτωρ Τσέγκερ, ήταν πάρα πολύ ε, δραστήριος και στρατευμένος και από τα 30-33 μέλη συγκεκριμένα ήταν ο μόνος ε, που αμφιταραντευόταν, ε, που ε, έκανε πάντα ε, ξεχωριστή δήλωση στην ψηφοφορία και κατέθεσε ξεχωριστή ψήφο. Σε ό,τι αφορά επίσης τη μείωση των συνεδριάσεων, αυτό είναι παραπληνητικό, γιατί το, συνεδριάς, το Συμβούλιο αυτό δεν συνεδριάζει μόνο σε Ολομέλεια, αλλά και σε ομάδες εργασίας πάντα μιλάω για το Συμβούλιο Προστασία ε, Προσωπικών Δεδομένων. Ήταν πάντα πολύ εντατική η δραστηριότητά μα και μην μετράτε μόνο τι ολομέλειε, αλλά και τι ομάδε εργασία. Γιατί η πραγματική δουλειά, ξέρετε, γίνεται στι ομάδε εργασία. Και εκεί ήταν δική μου πολιτική ότι όταν έβλεπα ότι δεν θα έχω ομόφωνες αποφάσεις στην Ολομέλεια, αν τα θέματα είναι τόσο περίπλοκα και τόσο ευαίσθητα όπως θέματα ασφαλείας. Η γνωμοδότηση για την, για την οδηγία συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είδα ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε έτσι σύντομα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το θέμα. Ε, είναι πάνω από 30 σελίδε η γνωμοδότησή μα, βέβαια καθυστερημένα κάπω ομολογώ, με μία εβδομάδα καθυστέρηση, ακριβώ γι' αυτό το λόγο, γιατί είδα ότι χρειάζομαι χρόνο σε ομάδα εργασία. Δεν μπορώ σε τρει ώρε να βγάλω αυτή την απόφαση. Ε, ε, ε κάναμε δύο ομάδε εργασία και μετά ομόφωνα γνωμοδοτήσαμε με πάρα πολύ λίγε μόνο επικριτικέ παρατηρήσει και πάλι του εκπροσώπου των πρασίνων. Δηλαδή, όταν το θέμα είναι ακαθόδε και ε, ρεπτό και ευαίσθητο ε, κάνω ομάδες εργασίας. Ε, δεν είναι τόσο πολιτικά φορτισμένες όσο η Ολομέλεια. Γίνονται οι συζητήσεις καλύτερα και τότε έρχονταν και δύο πράσινοι. Λοιπόν, μην κοιτάτε τις στατιστικές, δεν είναι πάντα το απάβγασμα της αληθείας. Για τις διευθύνσεις IP στο διαδίκτυο και τον εντοπισμό κάποιων κινητών τηλεφώνων. Το θέμα ήταν τι γίνεται σε επίγουσες περιπτώσεις και έκτακτες ανάγκες. Οι αρχές ασφαλείας μας μας είπαν με τρόπο αξιόπιστο ότι σε επίγουσες περιπτώσεις, σκεφτείτε ότι στην Αυστρία έχουμε και τις Άλπες, έτσι, και συχνά το χειμώνα γίνονται ε, δυστυχήματα και πρέπει να τρέξουν ε, ομάδες διάσωσης, ε, ορεινής διάσωσης και αυτοί θα πρέπει να εντοπίζουν Πού βρίσκονται τα κινητά. Λοιπόν, πού να βρεις δικαστή ε, και Σαββατοκύριακο. Και δεν προλαβαίνουμε. Είναι επίγουσα η κατάσταση για να χρειαστεί η έκδοση απόφασης. Και αυτά πάλι τα έχουν επικρίνει οι πράσινοι. Αλλά ε, στη Βουλή ψηφίστηκαν οι προτάσεις μας αυτές με συντριπτική πλειοψηφία. Χάουσερ. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέγκερ Μπάουερ, δεν είστε ανεξάρτητος, είστε ο υποψήφιος του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος. Και όπως γνωρίζετε και είναι πολύ μεγάλο το λόμπι της Γεωργίας αυτό το κόμμα. Είπατε ότι είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το ΔΕΚ κήρυξε απαράδοκτα ε, κάποια στοιχεία που δημοσιεύονται για εκείνους που λαμβάνουν ε, γεωργικές δαπάνες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωργικές επιδοτήσεις καλύτερα. Ε, συμφωνείτε εσείς σε ένα κοινό σύστημα προσωπικών δεδομένων στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κατονομάζονται και να δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Απάντηση σαφέστατη. Ε, ε, εγώ αναγνωρίζω και δέχομαι την απόφαση του ε, ΔΕΚ, του Δικαστηρίου. Κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ πολύ κύριε Βέγκεμπάουερ. Στην εισαγωγή σας, ρητά, Αναφερθήκατε στη διαφάνεια και είπατε πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης. Στην απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι το ελεκτικό συνέδριο πολύ συχνά αποσιωπεί τα ονόματα των κρατών μελών. Και χαίρομαι και το βρίσκω θετικό ότι έχετε αυτή την εμπειρία από τη χώρα σας που γνωρίζετε και το Ελεκτικό συνέδριο και την πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο τι θα κάνετε στο μέλλον, πώς, πώς βλέπετε ε, την αύξηση της διαφάνειας και στον κατονομασμό των κρατών που έφτουν σε παρατυπίες. Στην γραπτή απάντηση απαντήσατε και για τον έλεγχο των επιδόσεων. Performance audit το λένε αυτό. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον με τις αιτήσεις εκθέσεις αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπετε να διαδραματίζει εκεί κανένα ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί αυτό είναι ο λογιστικός έλεγχος των επιδόσεων, αυτό είναι. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει ρόλο εκεί στον αυτοαξιολόγηση και αυτο έλεγχο. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση, για τη διαφάνεια. Ως προς τα ονόματα των κρατών μελών. Μα ακριβώς γιατί η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, αν καταφέραμε να δημιουργήσουμε εδώ περισσότερη διαφάνεια. Δηλαδή, για να μπορεί κανείς να διορθώνει τα κακό κείμενα, θα πρέπει να ξέρει ποια είναι αυτά τα κακό κείμενα. Και ε, θα με ενδιαφέρει και θα το καλωσόριζα να πήγαινα προς την κατεύθυνση αυτή. Έκανα όμως ε, και κάποιες συνομιλίες, ε, είχα επαφές με υπαλλήλους του Ελεκτικού συνεδρίου ε, που μου απάντησαν στην ερώτησή μου ότι αυτό θα σήμαινε, πώς να το πω, τεράστιες επιπλέον διοικητικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες ελέγχου και συλλογή στοιχείων. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, ότι θα ήταν στόχος και για μένα να εντοπίζουμε ακριβώς και για τις εργασίες, επαναλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ποιους τομείς χωλαίνουν ιδιαίτερα τα πράγματα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο ένα τομέα πολιτικής που ε, είναι στο επίκεντρο αυτό τον καιρό, αλλά θα με ενδιαφέρει να βολιδοσκοπήσω και τι γίνεται στη διοίκηση ε, του Ελεκτικού συνεδρίου και αν υπάρχουν δυνατότητες από πλευράς προσωπικού. Τώρα, για τον έλεγχο των επιδόσεων και εξολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι ρόλο έχει εκεί να διαδραματίσει το Ελεκτικό συνέδριο. Αν μου επιτρέπετε να επεκταθώ. Εγώ προέρχομαι από ένα ελεγκτικό συνέδριο το οποίο έχει μια διαφορετική κουλτούρα ελεκτική από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το Αυστριακό Ελεκτικό Συνέδριο. Όπως σας είπα ε, και προηγουμένως, δεν είναι ο κρατικός λογιστής ή ο κρατικός ε, συμβολεογράφος με τη δήλωση αξιοπιστίας, ας πούμε, όπως είναι στην Ευρώπη. Βεβαίως η απαλλαγή είναι σημαντικό και η προετοιμασία της απαλλαγής για το κλείσιμο το λογαριασμό που περνάει από την κάτω βουλή γιατί η Άνω Βουλή δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες όταν είναι ε, ομοσπονδιακός ο προπολογισμός, λοιπόν η κάτω Βουλή τα αποφασίζει και ε, το ελεκτικό συνέδριο ασχολείται με τον έλεγχο της ε, σκοπιμότητας και της αποτελεσματικότητας και έχει κάπως διαφορετικό γνώμονα. Ε, τι μας ενδιαφέρει. το σύνομο βεβαίως και η αποτελεσματικότητα αλλά και οι οικονομίες στον προπολογισμό. Βέβαια το πρώτο είναι το σύνομο. Αυτό είναι η δήλωση εξοπιστίας, ας πούμε ε, που κυρίως εστιάζεται η Ευρώπη. Αλλά εμείς έχουμε αμέσως μετά την αποδοτικότητα ε, και ε, την αποτελεσματικότητα και αυτό είναι ο έλεγχο των επιδόσεων, αν θέλετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και το ελεκτικό συνέδριο να ε, προβληματίζεται για τη σκοπιμότητα, για το νόημα ορισμένων έργων, ορισμένων μέτρων και ορισμένων πολιτικών δράσεων σε τομείς πολιτικής. Και στη συνέχεια και τελευταία έχουμε την εξοικονόμηση πόρων, γιατί οι οικονομίες πολλές φορές δεν είναι ούτε σκόπιμες ούτε αποτελεσματικές. Ε, γι' αυτό είναι σε τρίτη μοίρα ε, το θέμα της εξοικονόμησης των πόρων. Και στο μέλλον, νομίζω και η κοινή γνώμη θα απαιτεί από το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό εννοώ, να εστιάζει περισσότερο στο βαθμό που γίνεται αυτό έτσι νομικά, σε αυτούς τους τομείς και να φύγει από τη δήλωση αξιοπιστίας και να περάσει και στον έλεγχο της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας και της ε, επίδοσης όπως το ονομάζουν τώρα στην Ευρώπη γιατί σίγουρα τα προγράμματα έχουν χώρο και η διοίκηση για μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα και καλύτερη λειτουργία. Ε, στο βαθμό που έχω την πολιτική αυτή δυνατότητα θα προσπαθήσω να το πράξω. Ευχαριστώ Κώστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω στην πρώτη απάντηση που δώσατε στην ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Και είπατε ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να αποδώσουν οι μεταρρυθμίσεις. Στο μέλλον πού βλέπετε ε, δυνατότητες να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ελεγκτικού συνεδρίου και να βελτιωθεί η λειτουργία του. Για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εδώ. Να μας πείτε πώς βλέπετε τη μελλοντική συνεργασία ελεγκτικού συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ε, επιτρέψτε μου να συνεχίσω εδώ αυτό ε, που απάντησα ήδη προηγουμένως ή άρχισα να απαντώ. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στο μέλλον του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση ακριβώς ελέγχου των οικονομικών, ελέγχου των επιδόσεων και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ε, το προσωπικό ε, πέρα από τη δήλωση αξιοπιστίας. Δηλαδή, χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των στελεχών, γιατί το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι υπόδειγμα στις οικονομίες, ε, στο προπολογισμό, θα πρέπει να αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και η πραγματογνωμοσύνη με αναδιάταξη των εργασιών και της λειτουργίας. Να στραφεί περισσότερο προς τη σκοπιμότητα, όπως σας είπα, και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας. Για να μπορεί το Κοινοβούλιο να συζητεί με λεπτομέρειες συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο ειδικών εκθέσεων. Έτσι, και κατά την άποψή μου θα πρέπει να αυξηθεί και η παραγωγή ειδικών εκθέσεων από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των δύο οργάνων, so, ich. πιστεύω ότι μπορώ να σας πω το εξής. Στο παρελθόν, επί σειρά δεκαετιών, Ε, Έλεγα λοιπόν, συγγνώμη, ε, στο παρελθόν, επί σειρά δεκαετιών, φρόντιζα ε, για αυτή τη συνεργασία. Ως ελεγκτής, όπως σας είπα στο ελεγκτικό συνέδριο, είχα πάντα εντατικές επαφές με τα κοινοβούλια, δηλαδή και με το Αυστριακό ε, Κοινοβούλιο, μας καλούσαν πάντα στις προπαρασκευαστικές τους ε, εργασίες ως ειδικού, ως εμπειρογνώμονες για να τους ενημερώνουμε. Βεβαίως πάντα με κάποιες δεσμεύσεις ε, απορρίτου και τα διάφορα νομικά που δεσμεύουν ε, τους υπαλλήλους. αλλά και στη συνέχεια στη Βουλή ως αρμόδιος για την Επιτροπή ε, ελεκτικού συνεδρίου καλούσα συναδέλφους από το ελεκτικό συνέδριο για να συζητούν μαζί μας και να προετοιμάζουμε τα πράγματα όχι μόνο στη δική μας πολιτική ομάδα, όλες οι πολιτικές ομάδες είχαν ίση μεταχείριση. Δεν πήγαιναν μόνο στα κυβερνητικά κόμματα ή σε κάποιες μόνο πολιτικές ομάδες ή πάλι του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό ήταν μια προσφορά εκ των προτέρων, επαναλαμβάνω, ε, προς όλες τις πολιτικές ομάδες για να έχουν πλήρη και ε, συνολική ενημέρωση με τους εκάστοτε ελεγκτές που ήξεραν και τα θέματα στις λεπτομέρειές τους. Και σε σχέση με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, εντείνεται κάτι τέτοιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι στη διάθεσή σας με μεγάλη χαρά να το πράξουμε. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βέκιο έχω δύο σύντομε ερωτήσει. Η πρώτη είναι κατανόηση, διευκρινιστική. Και η δεύτερη περισσότερο ουσιαστική. Στην υποψηφιότητά σας προς την ε, ε, Αυστριακή Καγκελαρία ε, να λέτε ότι είστε 36 χρόνια μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά βλέπω ότι επί μία πενταετία από το 1974 μέχρι το 1979 ήσασταν στο ελεκτικό συνέδριο και διατηρείτε αυτή την ιδιότητα. Εντάξει, δεν πειράζει αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα ε, και είπατε ότι ε, σας ενδιέφερε να παραμείνετε ε, κρατικός λειτουργός. Αυτό τι σημαίνει ότι από το 79 και μετά δεν έχετε ασκήσει καμία ουσιαστική ελεγκτική δραστηριότητα ως ελεγκτής του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή, το δεύτερο είναι θέμα ουσίες περισσότερο. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται με τον έλεγχο της εκτέλεσης του προπολογισμού και θέλει να είναι καθαρή η τήρηση ε, το λογαριασμό για να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι είναι κοινή η διαχείριση με τα κράτη-μέλη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχουμε την εμπειρία, πώς να το πω τώρα προσεκτικά, ότι δεν είναι συχνά ικανοποιητική η συνεργασία μας με τις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη που υποχρεούνται να δηλώνουν ε, ε, πώς γίνεται η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, δεν ε, δηλώνουν σωστά ε, όπως θα θέλαμε. Ψηφίσαμε την έκθεση του αδέλφου πρόσφατα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διαβάζω ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Αυστρίας ανήκει στα κράτη εκείνα που σε ό,τι αφορά τις παρατυπίες κυρίως στη Γεωργία και τις διάφορες ε, ατασταλίες δεν αναφέρουν, εν πάση περιπτώσει δεν αναφέρει η Αυστρία εγκαίρως αυτές τις καταστάσεις. Με βάση αυτά τα ευρήματα, πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα άσκηση και εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη συνθήκη για την Αυστρία, για ε, διαβίβαση και ενημέρωση και κοινοποίηση, εν πάση περιπτώσει, προ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα των καταστάσεων αυτών. Για την πρώτη σα ερώτηση, για το ελεκτικό συνέδριο και κατά πόσο συμμετέχω ακόμα εκεί. Σωστά παραθέσατε ότι ήμουν ελεκτής από το 74 έως το 79. Στη συνέχεια όμως δεν πήρα μετάταξη, αποσπασμένος είμαι. Δηλαδή, ε, παρέμενα υπάλληλο του ελεγκτικού συνεδρίου και διατηρούσα τα καθήκοντά μου και τις αρμοδιότητές μου και ε, ε, ήμουν αποχρωμένος να το πράττω αυτό και στα πλαίσια της πολιτικής μου δραστηριότητας. Επίσης ξέχασα να πω ότι ε, δεν ε, συμβούλευα μόνο την Επιτροπή του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και εξεταστικές επιτροπές. Και στις εξεταστικές επιτροπές πραγματικά μας ενδιαφέρει να ελέγχουμε την εκτέλεση των λογαριασμών, την, των προπολογισμών. Και εγώ ε, προετοίμαζα τις εργασίες και βεβαίως ήλεγχα ως οικονομικός ελεγκτής, ως επιθεωρητής λογαριασμών, γιατί ήταν αρμοδιότητά για τον κάθε τομέα ε, πολιτικής που χρειαζόταν. Αυτό ήταν ε, απάντηση στην πρώτη σας ερώτηση. Τώρα, κατά πόσο είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να ε, αναφέρουν πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τα όσα λέτε ότι ε, τα προβλήματα είναι μόνιμα και επαναλαμβανόμενα. Όταν η έκθεση δεν είναι έγκαιρη υπάρχουν τρόποι και μέσα ε, να επισημαίνεται αυτό πολιτικά και να επιβάλλεται και αν μπορώ να βοηθήσω σίγουρα θα το πράξω. <clears throat> Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε γιατί πρέπει να περάσουμε στην αξιολόγηση της ακρόασης και την ψηφοφορία. φω Σέντερ τελευταία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ήθελα γιατί στην πρώτη μου τοποθέτηση Αναφέρθηκα στα στοιχεία. Σας είπα όμως ότι θα ξαναζητήσω το λόγο για να μπω σε λεπτομέρειες, ε, στο περιεχόμενο και να διευρύνω σε κάποια θέματα που δεν έθιξαν οι συνάδελφοί μου. Και πάλι διευκρινιστικά, γιατί είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Δεν απαντήσατε σε μια από τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχω ένα δελτίο τύπου εδώ ε, από την κοινοβουλευτική πολιτική ομάδα του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος της 21ης 12ου του 2010, εσείς ως διευθυντής που ήσασταν τότε ορίζεστε υποψήφιος. Εσείς παραμένεστε σήμερα διευθυντής στην πολιτική αυτή ομάδα ή όχι, ή ε, παρετηθήκατε ή έχει τελειώσει αυτή σας η ιδιότητα και αν ναι πότε γιατί αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί εδώ βλέπω κάπως να συγχαίεται ε, ο πολιτικός σας ρόλος, που είναι θεμητός, αλλά ε, με, το διοικητικό, με το επαγγελματικό ως εμπειρογνώμων. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στο κοινοβούλιο μας η Πράσινη είναι μια πολιτική ομάδα και πρέπει να συνεργάζεται και με τους πρασίνους. Δηλαδή είναι σημαντικές οι ε, απόψεις και των πρασίνων βουλευτών όσο και των υπολείπων και είναι δουλειά μας να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτές τις ε, αντιλήψεις και απόψεις. Και τώρα, σε σχέση με την ερώτηση 9, και πάλι ίσως είναι θέμα μετάφρασης, αλλά συνήθως είναι καλές οι μεταφράσεις μας. Τι μας λέτε εκεί για το ελεκτικό συνέδριο, ότι χρησιμεύει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως αρχή χορήγησης απαλλαγής, ως αξιολόγηση. Μα τώρα βρισκόμαστε εν πλήρη συζητήση με το Συμβούλιο για το πώς αναγνωρίζουν το, και πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για την έγκριση των λογαριασμών. Δεν μπορεί το ελεκτικό συνέδριο να αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ως ισότιμους στη διαδικασία της απαλλαγής και δεν έχουν τον ίδιο ρόλο. Επίσης γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Πάγια και ιστορικά το Κοινοβούλιο ζητάει να μειωθεί ο αριθμός ε, των μελών του Ελεκτικού συνεδρίου που είναι 27 σήμερα, ένας από κάθε κράτο μέλος. Και αυτό έρχεται σε κάποια αντίφαση με το θέμα της ανεξαρτησίας, γιατί αν είναι ένας από κάθε κράτος μέλος, ε, δεν είναι και συλλογικό σώμα πάρα πολύ, ε, έχουν και τις εθνικές τους, αν θέλετε, ιδιομορφίες. Τι λέτε γι' αυτό, να μειωθεί ο ρυθμός στο μελών του ελεκτικού συνεδρίου για να είναι πιο αποτελεσματική η εργασία του. Και επίση, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται λόγο τώρα για το επιτρεπό επίπεδο σφάλματο. Αυτό είναι ένα όρο, μια έννοια τη ε, επαγγελματική ε, λογιστική ε, οικονομικού ελέγχου. Και μια τελευταία ερώτηση. Ξέρετε ότι στη φετινή έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Απαλλαγή του 2009 η Αυστρία εμφανίζεται ε, ε, με υψηλό επίπεδο υποψίας απάτης για προς τους ιδίους πόρους. Τι λέτε για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Πολιτικός Διευθυντής, ναι, Συμφώνησα με τον εργοδότη μου αν ε, διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να ε, παρετηθώ από τη σημερινή μου θέση. Προφανώς θα παρετηθώ και από σύμβουλο του Κοινοβουλίου και θα επανέλθω πλήρως στην ιδιότητά μου του υπαλλήλου του Ελεκτικού συνεδρίου ως αποσπασμένος. Δηλαδή θα εγκαταλείψω και θα παραιτηθώ από στις πολιτικές μου θέσεις. Έχω παραιτηθεί ήδη, έχω παραιτηθεί από ε, μέλος της Επιτροπής για την εξασφάλιση των συντάξεων, από πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων και από άλλες θέσεις πολιτικές που κατήχα. Παραιτήθηκα από όλα αυτά τα αξιώματα. Ε, Βεβαίως, ε, αγνώντας την απόφασή σας, ε, δεν έχω ακόμα παραιτηθεί από την υπηρεσία μου, ε, από τον εργοδότη μου. Έχω μια σύμβαση με το κόμμα, με την πολιτική ομάδα του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος. Σε περίπτωση που με έγκρινεται θα διακοπεί αυτή η σχέση μου. Η απαλλαγή δίνεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Βεβαίως τον, τον αποφασιστικό λόγο έχει ε, το Κοινοβούλιο και την τελευταία λέξη κατόπιν ε, προτάσεως του Συμβουλίου. Στο δικό μας σύνταγμα είναι πολύ πιο αυστηρό. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι υποβοηθητικό όργανο της κάτω βουλής και ε, έτσι το αντιλαμβάνεται και η Αυστρία λόγω του συντάγματός της. Βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομικά δεν είναι τόσο πολύ κατοχυρωμένο αυτό. Η μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου και μείωση των μελών μπορώ να φανταστώ ότι γίνονται συζητήσεις εδώ για αυτή την αρχιτεκτονική του Ελεκτικού συνεδρίου από πλευράς Κοινοβουλίου, ενδεχομένω και Συμβουλίου, αλλά αυτό τον καιρό έχει οριστεί έτσι στις συνθήκες. Δική σας ε, αρμοδιότητα και καθήκον ε, το αλλάξετε αν θέλετε και να, αναλάβετε τις, ή να μην αναλάβετε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το επιτρεπτό ή αποδεκτό επίπεδο σφάλματος και ότι είναι πολύ ψηλό για την Αυστρία. Λαμβάνω γνώση αυτό, το σημειώνω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιωθεί. Περισσότερο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω επ' αυτού. Δεν είχα την ε, δυνατότητα ακόμα να επέμβω και να έχω καμία επιρροή σχετικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φόκεν Μπάουερ. Τώρα θα κάνουμε την αξιολόγηση με συνεδρίες και κλεισμένων του θηρών και μετά με σκύψη ψηφοφορία.